να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα που είναι τόσο κοντά σε εμά τους Ευρωπαίους και να δείξουμε και την αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Χάμς, ακολουθεί για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ο κύριος Κόβαλ. 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ